Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Mr. Bill, can have ε, και κύριοι, έχω την ιδιαίτερη χαρά να ε, σας ανακοινώσω ότι παρευρίσκεται ο Υπουργό Εξωτερικών κ. Καρλ Μπίλτ για να συζητήσουμε μαζί την εξωτερική πολιτική της Ένωση και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη. Και από εκεί και πέρα ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία του και να συζητήσουμε μαζί του και άλλα θέματα. Όπως ε, τι έγινε στη συνάντηση για τη Συρία, θέματα που έχουν να κάνουν με τους υδατίνους πόρους, με την παιδεία. Έχουν ε, σχέση με την ειρήνη ευρύτερα αυτά τα θέματα. Αλλά επίσης και ε, τι γίνεται με την ανάπτυξη, με τις εξελίξεις ή τις αρνητικές εξελίξεις της δημοκρατίας και κράτους δικαιού στις ε, νότιες γειτονίες και ανατολικής γειτονίας χώρες. Και χαίρομαι που έχει την ευκαιρία συζητήσει μαζί μας αυτά τα θέματα. Καλ, γνωρίζεις ότι την περασμένη εβδομάδα ε, ψηφίσαμε την ετήσια έκθεση για την ε, ΚΕΠΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί να μας βοηθήσει και στη συζήτηση. Δεν είναι ένα θέμα, ε, μόνο συγκεκριμένα που μας απασχολεί. Χρειάζεται ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη και ευχαριστούμε που βρήκε στον χρόνο να έρθει Το λόγο έχει ο Υπουργό Εξωτερικών τη Σουηδία. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Έλμαρ. Πάντοτε χαίρομαι όταν έρχομαι στο Κοινοβούλιο. Σήμερα έρχομαι διότι θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο για την ε, ίδρυση αυτού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε και μια ευρύτερη συζήτηση. Θα πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι εντάσσεται αυτή η ιδέα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στο γενικότερο πλαίσιο των δράσεών μας για να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βασικό παίκτη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της ειρήνης, Ξέρουμε ότι ε, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα και ε, η ιδέα για να αναδειχθεί σε βασικό παίκτη της ε, Διεθνού κοινή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γεννήθηκε ε, χτε. Ε, βήμα προ βήμα, σταδιακά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο λοιπόν θα πρέπει να εγγραφεί στο γενικότερο πλαίσιο, στο γενικότερο οπλοστάσιο των μέσων που χρειαζόμαστε εμεί, οι Ευρωπαίοι για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μα και να προαγάγουμε τι αξίε μα εν γέννη στον κόσμο. Θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα για άλλα ζητήματα που ανέφερε ο Έλμαρ. Και τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα, παρεπιπτόντως, ε, αναφέρθηκαν στην έκθεση Μπρόκατς, δεν τη λένε. Πολύ καλό αυτό το έγγραφο. Πολύ καλή σύνοψη, όχι μόνο των απόψεών σας, αυτό εννοείται, αλλά και των διαφόρων προκλήσεων που ε, θα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ε, διάφορα σχέδια ψηφίσματος και εκθέσεων μας φαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα, όπως παραδείγματος χάρη ε, ε, η γνωμοδότηση για τις ελευθερίες του διαδικτύου, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Άλλη έκθεση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία θα έχει αυτό το ζήτημα. Η έκθεση για την και πάει για τα ζητήματα ευρωπαϊκής Ασφάλεια και άμυνας, ε, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ε, θα έχουν ε, ιδιαίτερη σημασία. Στον Σμιτ, στην σύσκεψη, ω συνήθω κάναμε μια πάρα πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, στη σύσκεψη αυτή ανασχολήθηκαν και με κάποια οριζόντια ζητήματα που λησμονούμε ορισμένες φορές. Ε, κάνουμε γεωγραφικού χαρακτήρα συζητήσεις. Να, ένα πρόβλημα εκεί, ένα άλλο πρόβλημα παρακάτω. Όμως η οριζόντια προσέγγιση και τα οριζόντια ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όπως οι ελευθερίες στο διαδίκτυο. Είναι ένα εγκάρσιο ζήτημα που επηρεάζει πληθώρα άλλων ζητημάτων. Το θέμα των υδάτινων πόρων, το θέμα ε, της ε, παιδείας και της εκπαίδευσης ε, και πώς ε, σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά είχαμε μια συζήτηση για τη Συρία, για το τι μπορούμε να κάνουμε στη χώρα αυτή. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις ε, για τους Ευρωπαίους ε, τη σήμερα ε, ημέρα και μεγάλες προκλήσεις για τους πολιτικούς, για τους διπλωμάτες. Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό η ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό απηχεί και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αλλά σχετίζεται και με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ήπια ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία στο εγχείρημά μας να προωθήσουμε την ειρήνη αλλά και την ευμάρεια. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, όπως ε, ε, είπε ο Κλίντον στην εκστρατεία του, η οικονομία είναι ανόητη, αυτή έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να αρχίσει να λειτουργεί και πάλι η οικονομία, να χρησιμοποιήσουμε το μαγνητισμό, την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις κοντινές γειτονικές χώρες αλλά και τις πιο απομακρυσμένες για να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή. Οι πολιτικές που ακολουθούμε ε, στις γειτονικές μας χώρες ε, έχουν ιδιαίτερη σημασία και μπορούμε να είμαστε ε, αποτελεσματικοί στην δράση μας και να αποκτήσουμε αξιοπιστία στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Πώς να είστε αξιόπιστος στις πιο απομακρυσμένες περιοχές όταν στη γειτονιά σας δεν τα καταφέρνετε. Ε, ο Έλμαρ και εγώ ε, ήμασταν με τον Στέφαν Φίλε στην Ουκρανία πρόσφατα και συνεχίσαμε ε, να καταβάλουμε τις προσπάθειές μας για αυτή τη χώρα με στόχο την ανάπτυξη Είχαμε διάφορες ε, συσκέψεις ε, με τον ε, Επίτροπο Στέφαν Φίλε, με τον Έλμαρ. Δεν ξέρω εσείς αν το δέχεστε, αλλά ισχυρίζεται αυτό σε κάτι τέτοιες συσκέψεις ότι εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο. Εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι εκπροσωπώ το Συμβούλιο, αλλά μέλος είμαι του Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση. Ε, ε, και λιγότερο σε εκπρόσωποι των τριών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουμε κοινέ συσκέψεις με τον πρόεδρο Γιαννουκόβης παραδείγματο χάρη, δύσκολες συνεδριάσεις ε, με ξεκάθαρες θέσεις εμφωτέρων των πλευρών και το αποτέλεσμα αυτών των συσκέψεων μας προσδίδει την αξιοπιστία. Δηλαδή τώρα το αν θα επηρεάσουμε όντω την κατάσταση η ιστορία θα δείξει. Έχουμε πολύ σημαντικές εκλογές ε, στην Λευκορωσία, όσον νούπο. Θα δούμε αν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες οι εκλογές. Αν κάποιος το πιστεύει να σηκώσει το χέρι του, δεν βλέπω να σηκώνει κανείς το χέρι του. Αλλά πόσο άσχημη θα είναι η κατάσταση τελικά, είναι απογοητευτικά τα πράγματα. Προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις με διαφόρους τρόπους. Στη Γεωργία θα γίνουν εκλογές την 1η Οκτωβρίου. Ε, όταν ήμουν εκεί τις προάλλες ε, με το, ε, τον Πολωνό υπέξε συνειδητοποιήσαμε ε, ε, όλες τις δυσκολίες. Θα είναι η καλύτερη μέχρι τούδε εκλογική διαδικασία και μην ξεχνάτε ότι είμαστε στον Κάφκασο, αλλά ε, σταδιακά βελτιώνονται τα πράγματα γιατί έχουμε πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις σε σχέση με ε, τον διεκδικητή των εκλογών ε, που η προσωπική του περιουσία αντιστοιχεί στο ίμιση του ΑΕΠ της Γεωργίας. Ε, καταλαβαίνετε πόσο επίμαχα ζητήματα προκύπτουν από αυτή και μόνο την κατάσταση. Πάνω από 2.000 παρατηρητές θα έχουμε στην Γεωργία, ούτως ώστε να αποτιμήσουμε την ποιότητα της εκλογικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, 28 Οκτωβρίου, έχουμε τη σημαντικότητα τη εκλογική διαδικασία στην Ουκρανία ε, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν ήμασταν εκεί. Ε, ε, εγώ, Έλμαρα, από το Κοινοβούλιο και Επίτροπος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλήσαμε για τις προσδοκίες μας. Ελπίζουμε ότι θα είναι ελεύθερες και δίκαιες οι εκλογές. Ετίθεται και ζήτημα ορισμού, βεβαίως. Ένας από τους βασικούς πολιτικούς ηθήνοντες έχει φυλακιστεί υπάρχει ζήτημα πολιτικής λογοδοσίας και ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές ε, θα έχει καταλητικό ρόλο για τις μελλοντικέ σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Έχουμε και το υπερχόμενο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και θα δούμε ε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στη συνέχεια προς Ανατολά σε Μολδαβία θα ήθελα να συγχαρώ τη χώρα διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολε οι συνθήκες. Παρόλα αυτά προωθούν τη μεταρρυθμιστική τους ευρωπαϊκή ατζέντα και πρέπει να τους υποστηρίξουμε στον υπόλοιπο Κάφκασο είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ε, ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν κλιμακώνεται η ένταση. Είναι σχετικά περιορισμένο ο ρόλο εκεί πέρα λόγω του Ναγκόνο Καραμπάχ και τη διαδικασία του Μίνσκ. Όμω ε, θα πρέπει να έχουμε πείγνωση τη κατάσταση. Και σε πιο κοντινές περιοχές έχουμε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα Βαλκάνια, η... προχωράει η διαδικασία της διεύρυνσης της Κροατίας, η, επικύρωση γίνεται από χώρα σε χώρα και η Σουηδική κυβέρνηση, απουσία μου, χάρη στην απουσία μου θα έλεγα, παρά την απουσία μου, ε, αποφάσισε να επικυρώσει, να υποβάλει συγγνώμη προς επικύρωση από το Κοινοβούλιο την ε, Συμφωνία Προσχώρησης της Κροατίας. Είναι εξαιρετικά ε, περίπλοκη η διαδικασία, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα ληφθεί η απόφαση στη Σουηδία και βλέπουμε ότι μία χώρα μετά την άλλη ολοκληρώνει τη διαδικασία επικύρωσης. Ελπίζουμε να συνεχιστεί. Για το, τα υπόλοιπα Βαλκάνια νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διακόψουμε τις σταδιακές προσπάθειες ε, μπορούμε να μιλήσουμε για τι λεπτομέρειε ποια βήματα πρέπει να κάνουμε, αλλά παρότι μπορεί να είναι μακρύ ο δρόμο για κάποιε από αυτέ τι χώρε. και έτσι θα είναι, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα ε, στη γεωπολιτική σκηνή. Το σημαντικό είναι να ε, συνεχίσουμε να κάνουμε τα βήματα για να υπάρχει αυτή η πορεία προ τα εμπρός. Σήμερα η ταχύτητα δεν είναι ο αποφασιστικό παράγοντας από πολιτική σκοπιά. Το σημαντικό είναι να συνεχίσει να κινείται το πράγμα διαρκώ να διατηρείται ένας ε, σταθερός ρυθμός και η ταχύτητα ε, θα συνδεθεί με τα ε, αποτελέσματα, τα επιτεύγματα κάθε χώρα Υπάρχουν και εγκάρσια ζητήματα, οι υποδομές στα Βαλκάνια. Αυτό αυξάνει τις εντάσεις. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ασχολείται περισσότερο με αυτό το ζήτημα με τρόπο ώστε να μπορέσουν αυτές οι χώρες από οικονομικής, ενεργειακής πλευράς και πλευράς μεταφορών να ολοκληρώσουν, να ενοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Έχουμε προκλήσεις του τύπου οργανωμένη εγκληματικότητα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αναπτύξουμε αποτελεσματικότερα εργαλεία για να βοηθήσουμε αυτού που όντω θέλουν να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα στι διάφορε χώρε να μπορέσουν να το κάνουν και γίνονται συζητήσει στο Συμβούλιο σε σχέση με την προϊούσα διαδικασία διεύρυνση ε, τη ε, Κροατία ε, σε σχέση με τα νομοθετήματα. Δηλαδή, εξετάζουμε επί χάρτου αν υπαρκούν αυτά που, έχουμε, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ή θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση και να προχωρήσουμε λόγω της κυρίας σημασίας του ζητήματος. Η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε βασικό εταίρο της Ένωσης από διάφορες πλευρές. Ε, είναι η πιο δυναμική ε, ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα και ως προς την εξωτερική πολιτική είναι πρώτης τάξης εταίρος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ΣΥΠΑ, για όλους και η διαδικασία προσχώρησης εντάσσεται σε αυτό το γενικό πλαίσιο σε ολόκληρη αυτή την γεωγραφική περιοχή ανάμεσα στο ε, Νείλο και στον Ινδόποταμό, ε, ε, έχουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα και υπάρχουν λόγια ανησυχίας. Η Αίγυπτος είναι η χώρα, πώς να το έλεγα, ότι είναι πηγή ανησυχίας. Είναι βέβαια, αλλά Υπάρχουν θετικά σημάδια ε, στις ε, Βρυξέλλες. Ε, είδαμε ότι προχωράει η σχέση συνεργασίας με την Αίγυπτο και θέλουμε να συνεχιστούν. Ελπίζουμε ότι συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι θα χρειαστούν οικονομική βοήθεια και υποστήριξη, με τρόπο ώστε να μπορέσουν να διεξαγάγουν και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είναι καταλητική σημασία, όχι μόνο για την Αίγυπτο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, διότι αν αυτοί δεν καταφέρουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα με τις δημογραφικές εξελίξεις της χώρας ε, θα περιπλακεί ε, ακόμη περισσότερο ε, η κατάσταση σε 5, 6, 7, 8 χρόνια. Έχουμε μια πολιτική δέσμευση, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η δέσμευσή μας για οικονομικά ζητήματα είναι εξίσου σημαντική. Με απασχολεί ιδιαίτερα το τέλμα ε, σε αυτό που ακόμη ονομάζουμε ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Η ε, ειρηνευτική διαδικασία, ε, δεν ξέρω, διαδικασία είναι και δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή. Ε, θα κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση, είναι σίγουρο και όσο περισσότερο συνεχίζει η κατάσταση ως έχει, οι λύσεις ε, θα δυσχεραίνουν όπως για την, το αν θα είναι ένα κράτος ε, ή όχι ε, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα περιπλέκεται περαιτέρω η διαδικασία η κάθε Άστον και το επιτελείο της ασχολούνται πισταμένα με την κατάσταση, αλλά δυστυχώ δεν είναι στο χέρι μας η Συρία. Ας το θέσω ήπια ή συνιστά μεγάλη πρόκληση ε, για την συνείδησή μας ε, με πολλούς τρόπους αλλά και για την πολιτική μας. Ε, τι έγινε στην Συρία. Όπως και σε άλλες χώρες της Μέσης ε, Ανατολής είναι θρησκευτικά, θρησκευτικής προέλευσης δικτατορικά ε, καθεστώτα. Πρόκειται για δικτατορικά καθεστώτα, συγγνώμη, λαϊκά και δημιουργούνται Ε, προβλήματα ε, υπάρχουν ε, κίνδυνοι λόγω του κατακαιρματισμού των θρησκευτικών κοινοτήτων από την ε, Βηρητό μέχρι ε, την Πάστρα στο Μπαχρέιν ε, υπάρχει το ίδιο φαινόμενο και θα μας απασχολήσει αυτή η κατάσταση για πολλά χρόνια. Τι κάνουμε με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν ηγετικό ρόλο για την βοήθεια προς τους πρόσφυγες, για τη βοήθεια προς τη Συρία, ώστε να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όταν δεν είναι πλέον υπό να, να, να, ξεφύγουν από τον έλεγχο τη κυβέρνηση κυβέρνηση, αλλά μην αρχίσουν ε, άτακτα να τρέχουν αριστερά και δεξιά. Για την πολιτική διαδικασία, γιατί υπάρχει, ο Κόφι Ανάν ε, απέτυχε διότι ε, ήταν διχασμένο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο κύριος Μπραχήμι κάνει τώρα τον πρώτο γύρο και θα τον συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Η αξιολόγηση του, δηλαδή αν εκείνος κρίνει ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική διαδικασία. Αυτό θα είναι κάτι ενθαρρυντικό για να αποφύγουμε ε, την ε, σφαγή, την εκατόμβη. Για την ευρύτερη περιοχή τώρα έχουμε θέμα ε, προσφύγων διότι δεν λειτουργούν πλέον οι οικονομίες. Έχουμε σοβαρότατες εντάσεις ανάμεσα στις ε, θρησκευτικέ ε, κοινότητες. Η συνεργασία με το Λίβανο είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι η πιο ευπαθής χώρα. Μην ξεχνάτε όμως και την Ιορδανία διότι φέρει ένα βαρύτατο άχθος αυτή η χώρα, το Ιράκ όπου βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται τους τελευταίους μήνες τα πολιτικά προβλήματα και επηρεάζεται η χώρα σε μεγάλο βαθμό από τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και φυσικά η Τουρκία που ε, θα πρέπει να λύσει το κομμάτι των προβλημάτων που τις αναλογεί. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν χρειάζεται τώρα να, κρηγορήσω. Ήθελα μόνο να πω ε, ότι Ε, όταν παρακολουθήσει κανείς ε, την Αμερικανική προεκλογική εκστρατεία και ε, δικαίως μπορώ να το καταλάβω η εκστρατεία ασχολείται μάλλον με τα οικονομικά ζητήματα Έχουμε όμως ε, ξεκάθαρα την εντύπωση ότι η όρεξη ε, των ΙΠΑ για ένα ενεργό ρόλο σε διάφορες περιοχές του κόσμου δεν είναι όπως το παρελθόν. Ε, κάποιοι καλωσορίζουν αυτή την τάση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος των ΙΠΑ. Όταν ε, κάποιοι, ή μάλλον η ικανότητα ή η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει σε, στις ιδιαίτερα σημαντικές ε, περιοχές ε, του πλανήτη αυξάνεται γιατί προωθούμε τα ευρωπαϊκά ενδιαφέροντα και αξίες και δείτε τι κάνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική. Το 2003, πριν από πολύ καιρό, λάβαμε μία απόφαση για την ε, στρατηγική άμυνα. Αλλά ε, καλό ήταν το έγγραφο, καλέ οι αποφάσει, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια. Χρειαζόμαστε μία νέα ε, στρατηγική ασφάλεια. Υπάρχει απροθυμία στο Συμβούλιο. Κάποιοι θεωρούν ότι παρά είναι περίπλοκα τα ζητήματα και ότι γίνεται χαμό. Και α το αφήσουμε καλύτερα. Η Σουηδία, η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία είπαν α ξεκινήσουμε μία νέα διαδικασία που θα είναι λίγο πιο ελεύθερη για γιατί δεν εντάσσεται ε, στο αυστηρό περιθώριο των θεσμικών ε, οργάνων. Α είναι ευρύτερη η πολιτική μα. Αυτέ οι τέσσερι χώρε λοιπόν θέλουν να συνεργαστούν μέχρι την επόμενη άνοιξη και να καταλήξουν σε ένα σχέδιο για μια ευρωπαϊκή παγκόσμια στρατηγική. Αυτό δεν καλύπτει μόνο τα θέματα ε, τη ασφάλεια. Είναι ο τρόπο διάδραση και ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε τι εξελίξει στον κόσμο με τα υφιστάμενα μέσα και τα μέσα που θα χρειαστούμε στο μέλλον. Στη συνέχεια την Άνοιξη θα πάρουμε αυτό το έγγραφο και θα το ενσωματώσουμε στην επίσημη διαδικασία. Δηλαδή, Κοινοβούλιο, ε, Συμβούλιο, Επιτροπή και άλλοι. Όταν φτάσουμε στο 2014 που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτος ε, και για το μέλλον των θεσμικών οργάνων έχουμε τις εκλογές στο Κοινοβούλιο, νέα πρόσωπα θα καταφτάσουν αλλά ε, είναι κέρια σημασία η χρονιά Ε, ε, γιατί τώρα ε, μπορούμε να αναρρώσουμε επιτέλους από αυτά που έγιναν στο Σαράγιο. Και 100 χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και χειροκροτήματα. Δεν συμβαίνει συχνά στην Επιτροπή μας αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι ατέλειωτος ο κατάλογος των ομιλητών, πάνω από 14. Και επιτρέψτε μου να σας προτείνω το εξής. Να κλείσουμε εδώ τον κατάλογο πρώτον και δεύτερον να είστε σύντομοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε 1,5 λεπτό στην αρχή και μετά να το μειώσουμε. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε και θέλουμε να ακούσουμε και απαντήσεις. Πρώτος ο κύριος Σαλαφράγκα. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίσατε, Υπουργέ Μπίλτ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σε τόσο καλή φόρμα. Γνωρίζετε άριστα τις εργασίες του Κοινοβουλίου, την έκθεση Μπρόκ ακόμα και τη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα. Είπατε ότι για να έχουμε αξιοπιστία στο εξωτερικό θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τις δικές μας ε, πρωτοβουλίες κοντά στα σύνορά μας και μιλήσατε για τη βόρεια ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα στείλουμε και στη Γεωργία αντιπροσωπεία και ξέρουμε όμως και την νότια μας διάσταση και την πολιτική γειτονία. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας για το εξής γεγονός. Γιατί αναφερθήκατε στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές και τι σημασία έχει η οικονομία. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε τις προάλλες στην Ολομέλη με την κυρία Άστον. Αν έχουμε αξιοπιστία, αν μπορούμε να έχουμε αξιοπιστία στην εξωτερική δράση της πολιτικής μας και της κοινή μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα σωστά. Προχθές μας είπε ο κύριος Μπαρόσο ότι στο G20 Ρώσοι και Κινέζοι μας έκαναν να κοκκινίζουμε γιατί δεν είμαστε σε θέση να λύνουμε τα δικά μας οικονομικά προβλήματα στην Ένωση. Γι' αυτό ερωτώ κύριε Βίλτ, Μπορεί να είμαστε ε, το πρώτο μπλοκ ε, ε, εισαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες ή το πρώτο μπλοκ εξαγωγών ή το πρώτο μπλοκ χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκεί δεν έχουμε αξιοπιστία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πήρατε τύφος πρωτοβουλίες για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και στείλατε και ε, σχετικά επιστολές. Εσείς ως μέλος του Συμβουλίου μπορείτε να κάνετε μια πρώτη αποτίμηση για τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γκόμες. Θα καλύψει το χαμένο χρόνο του κυρίου Σαλαφράγκα. Κύριε Μπίλτ, αναγνωρίζετε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από την οικονομία. Γιατί δεν κάνετε τίποτα για αυτήν την ε, ζούγκλα, την οικονομική και τους οικονομικούς παραδείσους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική πολιτική μας δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί με τους ε, στόχους. Και πώς θα γίνει κάτι τέτοιο εάν αυτές οι μαύρες τρύπες εξακολουθήσουν να υπάρχουν και εάν όλα τα χρήματα που έχουν παρανόμως κερδίσει οι δικτάτορες έρχονται στην Ευρώπη. Λυπηθήκατε είπατε για, την, ε, για το θάνατο του ηγέτη της Αιθιοπίας ε, του δικτατορά, αλλά και ευτυχώς βεβαίως ε, ελευθερώθηκαν και οι δύο Σουηδοί ε, δημοσιογράφοι. Αλλά τι κάνουμε για την απελευθέρωση των, Αιθιο... των Αιθιώπων φυλακισμένων. Τι κάνουμε γι' αυτό. Δεν είναι Ευρωπαίοι άρα δεν μας ενδιαφέρει. Τι κάνουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει συνολικός διάλογος στην Αιθιοπία. Δεν μας ενδιαφέρει επειδή είναι μακριά από μας. Ξέρουμε τα προβλήματα στη Συρία. Τι κάνουμε έτσι ώστε να πιέσουμε, να πιέσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας, να μειώσουμε την δυνατότητα βέτο αρνησικυρίας σε αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι κάνουμε γι' αυτό. Η συνείδησή μας δεν μιλάει για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Όγιουλαντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ απολύτω με την ε, αξιολόγηση που κάνατε όσον αφορά την θέση Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον ε, διαρκώ ε, εναλλασσόμενο κόσμο. Αναφερθήκατε στον Αγκόρνο Καραμπάχα και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά την άποψή μου είναι ακόμα πολύ περιορισμένος. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε πώς είναι δυνατόν να ε, ε, επανοργανώσουμε την θέση μας όσον αφορά ε, αυτή τη διαμάχη, γιατί πρέπει να επιληθεί. Ένα άλλο θέμα, ίσως να σας πληροφορήσω, αλλά και ταυτόχρονα να στήσω την στήριξη και την συνεργασία σας. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή μας εδώ ενέκρινε σύσταση σχετικά με την υπόθεση Σεργέη Μαγνίτσκι και μάλιστα με μεγάλη ε, συνένεση ε, και πλειοψηφία εδώ ε, αποφάσισε η Επιτροπή μας να στείλει το θέμα στην Ολομέλεια. Βεβαίως γνωρίζετε στο Συμβούλιο το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Ευελπιστώ ότι εσείς και η κυβέρνησή σας θα στηρίξει την πρόταση αυτή έτσι ώστε να υπάρξουν κυρώσεις, άρνηση δηλαδή για θεωρήσεις ταξιδιού, ε, βίζες κτλ. για όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και ευρύτερα ε, να μας στηρίξει έτσι ώστε να μην δίνουμε άδεια ταξιδίου σε ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε θέματα διαφθοράς, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας, αλλιώς δεν θα προλάβουν να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Κυρία Μπράντνερ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπίλτε που είστε εδώ μαζί μα σήμερα. Πρωτού μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη. Δεν θέλω να πω κάτι για τη Λευκορωσία. Η αποστολή του ΟΑΣΕ είχε ε, δεν, δύο μέλη της αποστολής ΟΑΣΕ δεν μπόρεσαν να εισέλθουν. Η Μαρή Λουίζα Μπέγκα από τον Bundestag είναι και συνάδελφό μα. Δεν μπόρεσαν να, να, μπουν στη Λευκορωσία. Οπότε θα πρέπει να τονίζουμε ότι υπάρχουν και τέτοιου είδου προβλήματα. Θα ήθελα όμω τώρα να ασχοληθώ με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη που αναφέρατε. Νομίζω ότι ε, σε αυτή την περίοδο κρίσης, κυρίω οικονομικής κρίσης, πρέπει να ε, ε, ξεχνάμε συχνά πόσο σημαντικό σχέδιο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και σε ολόκληρη την Ήπειρο σημειώνονται ακόμη οι εξελίξεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι και θα έπρεπε να το προβάλλουμε στο εξωτερικό και να βοηθήσουμε όλους όσους αγωνίζονται για να επιτύχουν την ειρήνη ε, στη, στη χώρα τους, να τους βοηθήσουμε να ορθοποδήσουν ε, ε, ε, ε, βέβαια πρέπει να εξασφαλίσουμε τα απαιτούμενα μέσα αλλά και τη βούληση των πολιτών μας να εμπλακεί στρατιωτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Δηλαδή προτού επικρατήσει η βία σε μια κρίση να χειριζόμαστε την κατάσταση και στο κουτί εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εργαλεία Έχουμε και διάφορα άλλα διπλωματικά μέσα στη διάθεσή μας, ε, όμως υπάρχουν και μέσα που δεν έχει ακόμα στη διάθεσή της ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογος για τη διαμεσολάβηση, παραδείγματο χάρη, ε, επισήμως πως δεν γίνεται, διότι μιλάμε μόνο με, την, με μία πλευρά της σύραξης. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο ρόλος των αντιπροσώπων μας επιτόπου και ο τρίτος είναι η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από αντίστοιχε περιπτώσει. Ε, η κονδόμηση ενδογενών ικανοτήτων σε εκείνε τι χώρε από δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού είναι κλειδί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία ε, σε αυτέ τι χώρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Um, on the, on σε αυτό που μόλις είπατε συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό. Ε, βεβαίως θα δούμε πώς θα, δούμε πώς θα ε, μπούμε στις διάφορες ε, καταστάσεις αλλά το σημαντικότερο είναι να επεμβαίνουμε εκ των προτέρων έτσι ώστε να τις προλαμβάνουμε να ασκούμε τέτοια πολιτική έτσι ώστε να προλαμβάνονται αυτές οι κρίσεις και μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ένας ένα από τα συστατικά κομμάτια αυτής της μεγάλης εικόνας. Το να πηγαίνουμε, ε, βεβαίως ε, μας ενδιαφέρει να μπορούμε να πάμε και σε καταστάσεις ε, ακόμα και αν η διπλωματία έχει αποτύχει, ακόμα και αν είναι δύσκολο οι διπλωμάτες μας να πάνε σε αυτές τις χώρες. Μιλάμε για καταστάσεις όπου η ήπια δύναμη, η soft power της Ένωσης είναι ήπια μεν, αλλά εξακολουθεί να είναι δύναμη. Αυτή είναι η ιδέα, να έχουμε δηλαδή μία τάση συμφιλιωτική παντού σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την Ρωσία. Ε, έχετε πολύ επικεντρωθεί στην θέση Μαγνίτσκι ε, και πολύ καλά κάνετε, αλλά η μόνη επιφύλαξη που θα μπορούσα να έχω είναι να μην το στενέψετε πάρα πολύ, να μην δώσετε δηλαδή πολύ συσταλτική ε, ερμηνεία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήμουν προημερών στην ε, Μόσχα και ξέρω και τι είπε η Κάθη Άστον ε, στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια. Ήταν πολύ σαφής και πρέπει να σας πω ότι αυτό το ακούσανε στη Μόσχα. Ήταν προφανές. Ακούσανε όλο το μακροσκελές μήνυμά της. Τα νέα έκτοτη είναι ότι ε, η ομάδα αυτή έχει κλείσει τα γραφεία της ε, στη Μόσχα γιατί δεν φαίνεται ότι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι και πολύ ευπρόσδεκτη. Βλέπω και τον ε, Ναβάρνη και ξέρω ότι πάρα ότι εκκρεμούν εναντίον του πολλές κατηγορίες για φοροαποφυγή και για διαφθορά κτλ. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Η υπόθεση Μαγνίτσκι ολοκληρώθηκε τραγικά με ένα αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε. Ε, πρέπει να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους ε, που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Και εδώ επανέρχομαι πάλι στο soft power. Σχέση με την οικονομία, ναι, τι να σα πω, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σα πω, ε, μη με βάζετε δηλαδή να σα πω τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να τροποποιηθεί, να μεταρρυθμιστεί η οικονομία και η αντιμετώπιση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομία. Οικονομίας. Μιλάμε για την ευελιξία τη οικονομία μα, ε, ε, μιλάμε για μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστήματων, μιλάμε για ένα σώρο πράγματα, είναι τρομερό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε τώρα να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Αυτό που έλεγα το λέω με πολύ μεγάλη μετριοπάθεια και ταπεινοφροσύνη. Πριν από 20 χρόνια τα πράγματα ήταν διαφορετικά και μπορούσαμε να κάνουμε ε, διαφορετική πολιτική γιατί η οικονομία ήταν και διαφορετική. Αν δει κανεί, α πούμε, τι ε, χώρε τη ε, Βαλτική που έκαναν τρομερέ μεταρρυθμίσει, θα διαπιστώσει ότι τώρα πλέον βρίσκονται σε ανωδική πορεία. Άρα αυτό μπορεί να γίνει σε μεμονωμένε χώρε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αλληλεγγύη και είμαι, είμαι αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρουμε. Η οικονομία μας ε, ε, δείχνει έτσι λίγο άρρωστη και αυτό ίσως έχει ένα κακό αντίκτυπο στο, στην, ε, στην οικονομία. Αλλά μην ξεχνούμε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα από εμάς ε, βέβαια το πραγματικό ερώτημα για μένα είναι προς τα που πηγαίνει η κινέζικη οικονομία. Ε, γιατί για τις ΗΠΑ ξέρουμε ότι έχουν προβλήματα, έχουν ε, μεγάλα ποσοστά ελλείμματος κτλ. Τι θα γίνει, τι θα γίνει με την Κίνα προς τα που πηγαίνει. Επίσης τι θα γίνει με τη Ρωσία. Δεν είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αλλά πρέπει παρότι η Ρωσία έχει μεγάλη τεχνογνωσία, έχει απίστευτο δυναμικό σε κόσμο, σε μυαλά, σε εγκεφάλους, ε, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να διαφοροποιήσουν την ε, εξάρτησή τους από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Επομένως παραμένουν ανοιχτά πολύ ουσιώδη και κεντρικά ερωτήματα. Ας δούμε λοιπόν εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας ουσιώδη προβλήματα και ερωτήματα, ε, να δούμε πώς εμείς μπορούμε να κλείσουμε τα ελλείμματα τη οικονομία μας, πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την οικονομία μας και οι άλλοι α κάνουν αυτό που νομίζουν επίση. Και μπορεί κανεί να προσθέσει ότι αν καταφέρουμε να μεταρρυθμίσουμε την οικονομία, θα πάρει και κάποια χρόνια βέβαια αυτό, μετά φυσικά θα ε, ε, γίνει και πιο δυνατή, πιο έντονη, θα αυξηθεί αυτή η ήπια δύναμη που έχουμε, αυτή η soft power που έχουμε. Ε, υπάρχει ένα μοντέλο που λέει ότι αυτά που έκανε η Ευρώπη μέχρι τώρα ε, ε, ήταν πρότυπο για τον κόσμο. Άρα ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει και την κρίση θα αποτελέσει πρότυπο για τον κόσμο πάλι. Άρα πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Αιθιοπία. Κυρία Γκόμες. Αναφερθήκατε σε εξελίξεις τελευταίες στην Αιθιοπία. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη χώρα Περιπλοκική ιστορία της. Αλλά ενδεχομένως δεν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην ε, ε, Αφρική μετά την ε, Νιγηρία. Άρα δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Λέτε ότι χρειάζεται inclusive dialogue, διάλογος με όλους, συνολικός διάλογος. Ναι, συμφωνώ. Τώρα, μαζί με τους Αμερικανούς, μαζί με, άλλους, ε, με άλλες χώρες οι οποίες έχουν σχέση με την ε, Αιθιοπία, εγώ ασχολήθηκα μαζί με τον Λουί Μισελ, ε, συζητήσαμε για το θέμα αυτό. και με τον Σόντερς που θα είναι εδώ και σήμερα το απόγευμα ε, όλοι να συνεργαστούμε έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε και να βοηθήσουμε την ε, Αιθιοπία να πάει προς το σωστή κατεύθυνση όσον αφορά ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και, και αν εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό για τη χώρα. Κύριε Σαλαφράγκα, τι θα κάνουμε, πού βρίσκεται η γραμμή της Ευρώπης; Νομίζω ότι η οικονομική κρίση όντως έχει επηρεάσει την αξιοπιστία μας συνολικά. Ναι, υπάρχουν ε, κάποιες ε, καλές ε, επιτυχίες όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια αρνητικά. Τι να κάνουμε. Κάποιοι από τους συναδέλφους το έχουν κάνει και αυτοί όταν ας πούμε κάνουμε διμερή σχέση με το Πακιστάν, με το Αφγανιστάν. Εγώ ας πούμε εκτός από τον Σουηδό πρέσβη έχω και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητούμε ε, των Ηνωμένων Πολιτειών συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι. Υπάρχουν ε, μερικές χώρες που είναι πραγματικά μεγάλες χώρες, ε, ε, τουλάχιστον αυτό διατείνονται και οι ίδιες. Δεν θέλουν να παίρνουν τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και να, να ενδυναμώσουμε καλύτερα τη θέση μας. Τώρα, Μπορεί κανείς να πει ότι δεν κάνουμε αρκετά. Εγώ ας πούμε έχω πολλές ιδέες. Π.χ. να έχουμε έναν, ε, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο ε, Μόνιμο Συμβούλιο Ασφαλείας μεταξύ των μονίμων μελών. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει τώρα, προφανώς, αλλά θα ήταν η, το, το όνειρό μου ας πούμε. Αυτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η επόμενη. Και έχασα και τη λίστα μου. Ο κύριος Ντονζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε να ανταλλάξουμε απόψεις ε, με τόσο ειλικρινή τρόπο και τόσο ευρύ διάλογο πάντα είναι ε, πολύ ενδιαφέρον. Για το Ινστιτούτο ε, για την Ειρήνη εσείς και η Φρανσίσκα παρουσιάσετε αυτή την πρωτοβουλία και τη βλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον και συμπάθεια. Αλλά τι γίνεται με τον πολλαπλασιασμό των δομών και των θεσμών, όχι για αυτό το συγκεκριμένο. Ας πούμε αυτό που είπε ο κ. Σαλαφράνκα, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι μια ευρύτατη μηχανή, βαριά, που μου φαίνεται ότι γίνεται σιγά σιγά πολύ γραφειοκρατική, δύο χρόνια μετά τη έναρξη της, εγώ προβληματίζομαι για το πώς λειτουργεί, πώς έτσι προτεραιότητες. Αυτό το λέει και η έκθεση Μπροκ και πώς όλα αυτά εμείς τα συνδυάζουμε για να έχουμε μια ε, συνολική και παγκόσμια προσέγγιση, όπως λέει η κυρία Άστον. Έχουμε εργαλεία και μέσα, αλλά δεν εξαντλούμε τις δυνατότητες. Μήπως θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε αυτά με έτσι μια κρίσιμη ματιά, να δούμε τι εργαλεία έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, τα οποία είναι αναξιοποιητά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Ας πούμε, η ΕΠΑ ε, τα αμυντικά στοιχεία μπορεί να είναι μετριοπαθή, αλλά ε, υπάρχουν και υποχρησιμοποιούνται αυτό τον καιρό. Και άλλο ερώτημα για τη Γεωργία. Πήγατε με τον κύριο Σικόρσκι και στη Ρωσία λίγο αργότερα. Ε, υπάρχει εκεί μια αποστολή δική μας που λειτουργεί πολύ καλά, δουλεύει πολύ καλά, η UMM, αλλά οι Ρώσοι δεν συμφωνούν να πάμε από την άλλη πλευρά των διοικητικών συνόρων με την Ασετία. Ε, τι έχετε να απαντήσει σε αυτό. Ευχαριστώ κύριο Κύριλοφ. Κύριε Μπίλτ, θέτω και πάλι το θέμα, γιατί δεν απαντήσατε. Ε, ε, σε σχέση με τις έντονες αψημαχίες Αζερβαϊτζάν, ε, Αρμενίας μετά την υποδοχή ε, ε, του Αζέρου αξιωματικού. Και τώρα αυτά επηρεάζουν τις πολιτικές. Ποιος πιστεύετε πρέπει, πρέπει να είναι ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση αυτής της κρίσης πέρα από το να προωθούμε τα όσα κάνουν άλλοι δύο μεσολαβητές του ΟΑΣΕ ε, δηλώνεται ότι ο ρόλος μας είναι πολύ περιορισμένος θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένος να ξεσπάσουν εκεί εχθροπραξίες θα είμαστε στην ίδια κατάσταση ε, όταν ξεκίνησαν τα πάντα μεταξύ Γεωργίας Ρωσίας και για το ορεινό Καραμπάχ πιθανότατα οι Ρώσοι να είναι ε, με την πλευρά των Αρμενίων και εμείς θα είμαστε με την πλευρά των Αζέρων και μία από τα ίδια. Λοιπόν, έχουμε ψηφίσματα και για τις δύο χώρες ε, που μιλούμε για τη συμφωνία σύνδεσης ε, της οποία συνδέουμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων με την ειρηνική επίλυση του ε, ζητήματος του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εμείς εκεί τι κάνουμε ως Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμστορφ. Uh, Ευχαριστώ. Ε, πάντα με χαρά σας ακούω σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη. Πρώτον, πώς θα εξασφαλίσετε την υποστήριξη των κρατών μελών. Ακούσατε από τον συνάδελφο Ντονζό ότι η γαλλική ε, θέση θα είναι πολύ επιφυλακτική για να το πω ήπια. Ξέρω Αρνό ότι δεν εκπροσωπείς εδώ τη γαλλική κυβέρνηση, αλλά έχουμε δει και τη γαλλική θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν ήθελαν ισχυρό ρόλο ε, για την υπηρεσία και την ΚΕΠΑ καθόλου και ήταν και κατά του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και πιθανότατα και κατά αυτού του Ινστιτούτου θα είναι η Γαλλία. Χρειάζεται νομίζω να πηγαίνετε λίγο περισσότερο στο Παρίσι ε, για να του πείθετε και λίγο εκεί. Λοιπόν, πώ θα εξασφαλίσετε την υποστήριξη, λέω, των κρατών μελών. Γιατί πραγματικά έχει μεγάλο νόημα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέσο, ένα εργαλείο πιο ευέλικτο, α πούμε, και μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και ένα δεύτερο. Πώ φαντάζεστε να διασυνδέεται αυτό με την υπηρεσία εξωτερική δράση. Αυτό το Ινστιτούτο, τι θα είναι. Ε, θα είναι κάτι τοπικό, ε, θα είναι τμήμα της ε, επίσημης δομής τη υπηρεσία εξωτερική δράση, Το έχετε σκεφτεί αυτό, σας προβληματίζει. Και πόθεν η χρηματοδότηση, αυτό το έχετε εξετάσει. Όχι, γιατί έχει έρθει η ώρα να μπούμε στα συγκεκριμένα. Γιατί το 2014 είναι σε 14-15 μήνε από σήμερα. Ε, όλους μαζί θα τους ομοδοποιήσουμε και μετά θα απαντήσετε. Η κυρία Μπριζάζης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάρλ, ευχαριστώ που σάρωσες όλο το πολιτικό πεδίο με στην παρουσίασή σου. Θα ήθελα δύο πράγματα μόνο να πω. Για την Κροατία θα γίνει προσχώρηση σύντομα ε, και παρόλα αυτά έχουμε τόσα εκρεμή ζητήματα ακόμη δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τις χώρες στη συνέχεια, δηλαδή μετά την προσχώρηση, αλλά ενώ παραμένουν τα προβλήματα. Τα ζητήματα ανάμεσα στην Κροατία και τη Βοσνία παραμένουν ακέραια. Και υπάρχουν πράγματα, προβλήματα θα έλεγα με άλλες γειτονικές χώρες της Κροατίας. Με ποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε επικοδομητικοί, Πώς μπορούμε να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να επιληθούν τα ζητήματα όχι μόνο πρώτης προσχώρησης αλλά και μετά την προσχώρηση της Κροατίας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, η κατάσταση που ζούμε σήμερα προσπαθούμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Έχουμε χώρες όπως η Λιθουανία, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει επικυρώσει τη Συμφωνία Σταθερότητας, ε, Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ε, με την Σερβία. Υπάρχουν και άλλες χώρες ε, που επίσης δεν την έχουν επικυρώσει. Τι συζητείτε τώρα στο Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα. Ε, συζητάτε εσείς διμερώς με τη Λιθουανία για να ασκήσετε πίεση και να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συμφωνία. Η κυρία Ρωμέρο Λόπες, καλά τι είπα κύριος, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπίλτ και να αναγνωρίσω το ρόλο που ανέκαθεν διαδραμάτιζε η Σουηδία ε, στον αγώνα για την ειρήνη. Θέλω να θυμίσω τον πρόεδρο Πάλμε ε, της κυβέρνησης της ε, Σουηδίας και όλα όσα έκανε. Αναφερθήκατε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εγώ να αναφερθώ στο δεύτερο και όλες τις συμβάσει τη Γενέβης που υπογράφησαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα τι γίνεται, πολλές χώρες ε, που είναι συμβαλόμενα μέρη δεν τις στηρούν. Υπάρχει λοιπόν ένα διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και σήμερα που γίνεται πόλεμο στη Συρία ε, βλέπει να μην ε, τηρούνται οι συμβάσεις για τους εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες, τον άμαχο πληθυσμό, ε, τα γυναικόπαιδα. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό. Ε, τι μηχανισμούς έχει η Ευρώπη για να μπορέσει να επιβάλλει την εφαρμογή τους. Τι θα κάνει στο Συμβούλιο η Σουηδία και το Ινστιτούτο για την Ειρήνη. Μιλούμε για πρόληψη, για αποτροπή, ε, όμως δεν μιλούμε η ήπια δύναμη δεν πρέπει να είναι ασθενής δύναμη και η αποτροπή είναι ο τρόπος που θα επιτύχουμε την ειρήνη. Ευχαριστώ. Yes, whatever means. Um, it is of course true that if all of the conventions... Ό,τι και αν σημαίνει αυτό βεβαίως, ε, νομίζω ότι ό,τι αποφασίζεται ε, ε, και για να επιτύχουμε την μάλλον ό,τι αποφασιστεί σημαίνει ότι ε, συμμόρφωση μόρφωση όλων ε, και ζούμε όλοι σε ένα ρόδινο κόσμο. Ξέρετε, ε, παραβιάζονται αυτές οι συμβάσεις σε διεθνείς συνθήκες ε, και γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Και δεν παραβιάζονται γιατί κάποιοι θέλουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους ή οτιδήποτε. Αλλά ε, στις διάφορες συνθήκες φαίνεται ένας ιδεαλισμός που έρχεται αντιμέτωπος με την ομή, σκληρή πραγματικότητα ε, στον πραγματικό κόσμο. Σταδιακά λοιπόν με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δώσουμε μία όθηση. Ε, διαβάζουμε βιβλία ιστορίας και ξέρουμε σε ποιο κόσμο ζούμε, ξέρουμε ότι δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη ε, αυτό που θέλουμε αλλά σταδιακά μπορούμε να βρούμε τρόπους για να επιτύχουμε αυτά που επιθυμούμε. Άννα μίλησες και σου ειδικά να το αναφέρω και αυτό. Το θέμα της ε, Λιθουανίας ε, δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχουν επικυρώσει τη συμφωνία. Ε, σε παρακαλώ να μου δώσεις περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι στα Βαλκάνια υπάρχουν διάφορα προβλήματα, μεγάλα και μικρά. αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που εκρεμεί ζητήματα ανάμεσα στην Βοσνία και την Κροατία. Ε, κάποτε ήταν μία χώρα όλες αυτές οι χώρες. Πριν από πολύ καιρό το διαβάσαμε στα βιβλία της ιστορίας. Τώρα όμως ε, υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στις ε, δύο χώρες. Και τα ε, σύνορα είναι κάτι αμετακίνητο. Από βοσνιακής πλευράς υπάρχει αντίσταση για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. και οι Βρυξέλλες ε, δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσα προβλήματα θα προκύψουν την 1η Ιουλίου για τους ε, μεθοριακούς ελέγχους, για τη γεωργία, για τους υδάτινους πόρους, ε, μία σειρά ζητημάτων που αφορούν πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε με τους ε, δύο υπουργούς εξωτερικών των χωρών αυτών της προάλλης της Βρυξέλλες και όντως πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά αυτές τις μάλλον τεχνικές συζητήσεις και όντως θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να επιληθούν αυτά τα ζητήματα και να μην επηρεαστεί αρνητικά η καθημερινή ζωή των ανθρώπων μετά την προσχώρηση. Κύριε Λάμστορφ, ε, αναφερθήκατε σε διάφορα ζητήματα. Θα απέφευγα να σας δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση τελική απάντηση για κάποια από αυτά. Ας δούμε τι θα γίνει. Αλλά ε, δεν θα ήθελα να δείτε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, ε, διότι αυτό έχει και κάποια μονεκτήματα ένας ανεξάρτητος θεσμός που βρίσκεται στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως να έχει μία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβουλίο, όμως να διατηρεί το περιθώριο ελιγμών και την ελευθερία κίνησης και να μην περιορίζεται από ε, την γραφειοκρατία. Ένας ανεξάρτητος οργανισμός ε, και φτάνουμε στο βασικό ζήτημα της χρηματοδότησης. Ε, ε, ενδέχεται να προκύψει χρηματοδότηση από κάποια κράτη-μέλη αλλά και από άλλα θεσμικά όργανα, δηλαδή μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα υποστηρίξουμε αυτό το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο, να βρούμε ένα μίξε χρηματοδότησης που να ακολουθεί την, το καθεστώς ε, την, ε, του οργανισμού, το ε, ανεξάρτητο ή μη ανεξάρτητο, την ή ανεξάρτητη υπόσταση του οργανισμού. Διότι εάν δεν έχει αυτή την υπόσταση, ίσως απολύσει και την ικανότητά του να παρεμβαίνει. Δηλαδή, προσπαθήσουμε να μεθοδεύσουμε μία λύση που θα καλύπτει όλες αυτές ε, τις πτυχές. Ε, ε, θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας να πηγαίνω συχνότερα στο Παρίσι. Δεν μπορεί να έχετε και άδικο. Θα δούμε τι θα κάνει η Γαλλία. Για τον Αγκόρνο Καραμπάχ και το Αζερμπαϊτζάν. Ε, πολλοί θα το ήθελα να είχαμε ενεργότερο ρόλο, αλλά δεν έχουμε. Προσπαθήσαμε και στην Σουηδική Προεδρία να καταλήξουμε ε, σε μια ελάχιστη ε, ευρωπαϊκή θέση. Ε, και κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να μπλεχτούμε σε μια διαδικασία που ε, εμφάνιζε κάποια σημάδια προόδου. Ε, στη, με την ανατολική εταιρική σχέση και την πολιτική ε, ανατολικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καταφέρουμε κάποια πράγματα και μπορεί με την Αρμενία να θεωρείται ότι έχουμε ικανότητα επιρροή, Υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης, αλλά Πρέπει να προσέξουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε και να αντλήσουμε τα διδάγματα από αυτά που συνέβησαν το 2008. Δηλαδή, αγνοήσαμε τα σημάδια του επικείμενου πολέμου, κοιτάζαμε προς μία άλλη κατεύθυνση και ξέσπασε ο πόλεμος ε, ξαφνικά και αυτό μπορεί να ξανασυμβεί ε, σε αυτήν ε, την περιοχή του κόσμου και εμείς θα πρέπει να είμαστε ε, καθόλου προετοιμασμένοι για να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη στη ρίζα της. Ε, εάν εξεσπάσει πόλεμο στον Αγκόνο Καραμπάχα από το Ιράν μέχρι τη Ρωσία θα δημιουργηθούν σοβαρότατες εντάσεις και μπορεί να είναι βαθύτατες οι επιπτώσεις μιας τέτοιας ένοπλης σύραξης. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αξιολογούμε διαρκώς την ρόλο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Μπορούμε να πούμε πολλά θετικά πράγματα για την υπηρεσία. Αυτό που με εξέπληξε προσωπικά είναι το εξή. Ε, υποτίθεται ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα οδηγούσε σε μια καταπληκτική αρμονία και συνδυασμό ε, όλων αυτών των πραγμάτων ίσως ήταν αφέλες γιατί πάντοτε υπάρχει, ε, ακόμη υπάρχει ένταση ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κάθε είναι και Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συνδέεται η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μάλλον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική γειτονία και τη διεύρυνση αυτό λειτουργήσε αισίως. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε διαφορετικού τομεί. αλλά τώρα το, το θέμα είναι να ολοκληρωθούν, να ενοποιηθούν αυτέ οι προσπάθειε, όπω σα είπα για την παγκόσμια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι μάλλον αμφίβολο για να είμαι και διπλωμάτης ε, και να χρησιμοποιώ ε, την διπλωματική γλώσσα όπως και εσείς. Είναι αμφίβολο λοιπόν αν θα, καταφέρει, θα το καταφέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πάντω σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μάθουμε ο ένα από τον άλλο. Κανεί δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Όταν του χρόνου αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για την υπηρεσία εξωτερική δράση, σίγουρα θα υπάρξει νέα έκθεση Μπροκ ή άλλη έκθεση από κάποιον άλλον. Σα άρεσε αυτό που είχα πει για την έκθεση Μπροκ. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η έκθεση θα ε, συμβάλλει σημαντικά στην ε, συζήτηση και από πλευρά Συμβουλίου Κρατών Μελών αποσκοπούμε σε κάτι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συγκρότηση ενός ε, τέτοιου οργανού όπως η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, έχουν γίνει ήδη πάρα πολλά πράγματα, αλλά ε, πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμη. Η Γεωργία, δεν αν το ανέφερα όταν πήγα στη Μόσχα, όχι, αλλά το έχω κάνει στο παρελθόν. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για την Γεωργία, ούτως ή άλλως ε, είναι μόνιμο ζήτημα στην ημερησία διάταξη όταν επισκεπτόμαστε τη Μόσχα, ε, αλλά ε, δεν ασχοληθήκαμε ειδικά με αυτό. Η UMM είναι πολύ σημαντική αποστολή της Ένωσης, χωρίς την παρουσία της Ένωσης θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο μέρος ο Κάφκασος σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Ξέρε, και δεν ακούμε πολλά πράγματα για την EUMM ακριβώς επειδή είναι επιτυχής. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, για τη Γεωργία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δώσαμε ουσιαστικότατη οικονομική βοήθεια μετά τον πόλεμο και σταθεροποιήθηκε η χώρα. Ε, Έχουμε, οργανώσαμε αυτή την αποστολή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ανατολική γειτονία και η προοπτική διεύρυνση είναι σαν φάρο σαν αστέρι που οδηγεί τις ε, εξελίξεις ε, στη χώρα ε, και νομίζω ότι αυτό θα, θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει μια επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τις σχέσεις με τους Ρώσους, για την Απχαζία και την Νότια Οσετία και την αναγνώρισή τους ως ανεξάρτητα κράτη, κατάφεραν τελικά τι. Όχι. Η Ναγούρου, η Νικαράγουα, ποιος άλλος έχει αναγνωρίσει. Ε, τέλος πάντων, ε, βλέπετε πώς, τι καταπληκτική επιτυχία είχε η ρωσική εξωτερική πολιτική. Τίποτα δεν κατάφεραν να κάνουν και ε, θα πρέπει ε, ε, σύν το χρόνο να έχουμε υπομονή και να αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θα συμβούν αυτά άμεσα. Θα αλλάξει η συναστρία, σας το λέω, στο μέλλον και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Και για την Απχαζία και για την Νότια Οσετία. να, συγκεκριμένα παραδείγματα όπου ε, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, όπου δεν λειτουργούν ε, τόσο πολύ άλλα εργαλεία. Είδαμε ότι η Ναχούρου έχει τα χρώματα της δικής σας ημέρας, γαλάζιο και κίτρινο. Α, τι να κάνουμε, δείξτε τα στους Ουκρανούς. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπουργέ. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ ενώπιόν μας. Ξανά και συμφωνώ με τα γενικά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις για τα Βαλκάνια. Γνωρίζετε ότι εδώ είμαστε πολύ ε, εκείνοι που νιώθουμε απογοήτευση για την κατάσταση σε κάποια κράτη των Βαλκανίων και τη Βοσνία ε, Ζεκοβίνη κυρίως, αλλά και τη Μακεδονία Φιρόμ, λέει κύριος Πέτερλε. Ε, θα ήταν ίσως χρήσιμο να δείξουμε μεγαλύτερη πολιτική φιλοδοξία σε σχέση με αυτά. Χρειάζονται βήματα πρόοδου, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ε, ενεχόμενοι σε αυτή την περιφέρεια, των οποίων τα συμφέροντα δεν εγγράφονται πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ούτε φυγραμμίζονται με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και περισσότερη Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να σημαίνει περισσότερη Ευρώπη στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και από ό,τι φαίνεται, τα Βαλκάνια ε, παραμένουν ένα τμήμα της ατζέντα για την ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να βοηθήσετε και να προσιλωθείτε και να αφοσιωθείτε. Και θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για τη Βοσνία, Ρεζεγοβίνη και τη Μακεδονία. Να μας πείτε τίποτα και για την Τουρκία. Ευχαριστώ. Και τώρα, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φουκλέος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίλτ για την παρουσίασή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τα όσα έχει πει. Περιορίζομαι στην αναφορά που έχει κάνει για την Τουρκία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι πρώτη τάξεως εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι θα εμπορούσε να είναι πρώτη τάξεως εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζει ο κύριος Μπίλτ ότι σήμερα συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία. Γνωρίζει ο κύριος Μπίρτ ότι σήμερα ακόμη συνεχίζει να μην αναγνωρίζει ουσιαστικά μια χώρα που είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι η σωρία ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή της Διεθνής Ένωμης Τάξης, ουσιαστικά δεν έγιναν αποδεχτά και σεβαστά από την Τουρκία και βεβαίως ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αν δεν αναγνώριζε την Σουηδία θα έλεγε τα ίδια ο κύριος Μπίλτ. Αν δεν άφηνε τα πλοία να λιμενίζονται στην Σουηδία ή σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, θα λέγατε τα ίδια. Και θέλω να κλείσω με μια θέση σαφή και ξεκάθαρη. Αναγνωρίζω κατά απόλυτον τρόπο, ξεκάθαρο τρόπο, ότι ο Σουηδικός λαός έχει προσφέρει πολλά για την ειρήνη και την νομιμότητα παγκόσμια. Ευχαριστώ. Dank. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, Ω ε, εισηγητή τη έκθεση για τη Γεωργία θέλω να σα ρωτήσω, μάλλον είχα την πρόθεση να σα ρωτήσω για τη Γεωργία και ε, απαντήσατε, οπότε δεν θα επαναλάβω. Έγινε μια ερώτηση για τη Γεωργία και για τον Αγκόνο Καραμπάχ. Ε, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και για την υπερδυνιστερία. Ε, και για να τα συνοψίσουμε όλα αυτά τα θέματα, από ό,τι φαίνεται, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δίνουμε την εντύπωση ε, ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα επικοινωνίας με τους εταίρους μας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ σε αυτή την υπόθεση, διότι το κλειδί για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι στη Μόσχα. Πώς θα πρέπει να επικοινωνούμε με τη Ρωσική Ομοσπονδία για να τους πείσουμε και να αναγνωρίσουν τα δικά μας επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσπέργης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ ε, που ήρθατε. Εγώ έχω μια μικρή ερώτηση. Γεωργία, 1η Οκτωβρίου. Συγκεντρώνονται στρατεύματα στα σύνορα ε, με τη Γεωργία σε προ, ε, ηγουμένως κατεχόμενες περιοχές. Θα συνεχιστεί η εισβολή. Μπορεί να βρουν μια πρόφαση, όπως έγινε και το 2008. που μπορεί να κάνει την κατάσταση έκρυφμη στις εκλογές. Και οι γεωργιανές ε, αρχές ίσως ε, αναγκαστούν να αναβάλουν τις ε, εκλογές κατά ένα μήνα ή δύο μέχρι να τελειώσουν οι στρατιωτικές ασκήσεις των Ρώσων εκεί στα σύνορα. Θα γίνει κάτι τέτοιο, λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Εάν καταφέρουν οι Ρώσοι ολιγάρχες να όρος ο ολιγάρχης μάλλον να κερδίσει ψήφους αρκετούς και να δημιουργήσει και ταραχές και διαμαρτυρίες γιατί να μην κερδίσει και αυτός και τα λεφτά του τις, οι εκλογές. Οι Ρώσοι που κάνουν γυμνάσια εκεί και κάνουν ασκήσεις μήπως πάνε και στην Τυφλίδα να κάνουν στρατιωτικές ασκήσεις. Μπορείτε να ρωτήσετε το Κρεμλίνο εκ των προτέρων τις προθέσεις του για να το βολιδοσκοπήσετε. Και μία δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η απόψή σας για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν τα θεσμικά ε, όργανα, για να μην μιλήσω για τις άλλες διαπραγματεύσεις που ναυάγησαν, ε, για ε, τη συζήτηση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ του Αζερπαϊτζάν που είναι υπό ε, ε, στρατιωτικό έλεγχο της Αρμενίας. Γιατί δεν θεωρείται εμπόδιο αυτό στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και γειτονικά εδάφη ε, γύρω από το Ζεπαϊτζάν που αργότερα ήταν υποκατοχή δεν φαίνονται ως πρόβλημα. Φαίνεται ότι η Ρώσο-Αρμενική Συμμαχία ε, θεωρείται ανωτέρα βία και κερδίζει έδαφος αυτή η άποψη στους διπλωματικούς κύκλους και σε διάφορες πρωτεύουσε για να ε, διαιωνιστεί αυτό το στρεβλό στάτους κβό. Αν δεν γίνει τίποτα ε, θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρήνη ε, θα είχε διαφορετική στάση, έτσι πιο επικοδομητική και καρποφόρα. Ευχαριστώ. Thank you very much, ε, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Όπως βλέπετε είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σας βλέπουμε και σας ακούμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι καλό ε, που ο κύριος Μπέρκης ρώτησε για τη Γεωργία, έτσι δεν χρειάζεται να το ρωτήσω και εγώ. Αλλά να πω το εξής, ε, ε, βλέπουμε πολλές προκλήσεις στη Γεωργία από τον κύριο Ιβανισβίλη, από την, πολλές προκλήσεις λοιπόν από την αντιπολίτευση και πολλοί πιστεύουν ότι είναι δάκτυλος της Μόσχας. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση εκεί. Δεύτερη παρατήρηση τον Αγκόρνο Καραμπάχα. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή εάν μου λέγατε πώς, ότι έχετε τη λύση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να ε, διευρύνετε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά. Να μην περιμένουμε να ξαναδούμε τα όσα συνέβησαν το 2008 στη Γεωργία, αν και πιστεύω ότι αν ξεσπάσει η πραγματική σύρεξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ θα είναι πολύ πιο σοβαρή. Είμαι Λετωνή και θα σας ρωτήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας. Οι ενέργειες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στην Gazprom ε, και δεν έχουμε πληροφορίες για αυτές τις έρευνες. Πώς βλέπετε την διαδικασία αυτή, έχετε κάποια άποψη για το πώς θα προωθηθεί η διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Ο Καρλ. Αυτή uh, τη τελευταία ερώτηση. Βέβαια αυτή τη διαδικασία την έχει εκκίνησει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των νομικών αρμοδιοτήτων της ε, και υποθέτω ότι ανησύχησε, εκνευρίστηκε στη Ρωσία η Γκάσπρομ και ζήτησε να μπροκαριστεί ενημέρωση. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά. Και γιατί να γνωρίζω. Άλλωστε, διότι είναι ανεξάρτητη αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε το Κοινοβούλιο ενημερώνεται, ούτε τα κράτη-μέλη. Στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε αποφασιστικότητα σε τέτοιες περιπτώσεις και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει την ίδια στάση και συμπεριφορά και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Για τη Γεωργία και αυτό που ρώτησε ο κύριος Λάσπεργης, πολλές ερωτήσεις μου κάνατε. Θεωρώ απολύτως ουσιώδες να πούμε ότι ε, ε, προς πάντα ενδιαφερόμενο ότι όλοι έχουν το χρέος να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού των ε, εκλογών και είναι πολλοί οι παρατηρητές, ε, πολύ περισσότεροι των εκλογών από οποιασδήποτε άλλες εκλογές και θα κάνουν την αξιολόγηση και την εκτίμησή τους την ίδια μέρα, την επομένη, τη μεθεπομένη, οπότε την κάνουν. Και αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει όλοι να το μελετήσουμε. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα, λοιπόν, σαφέστατα από πλευρά μου και προς τη Γεωργία την ίδια και με τη σημερινή πλειοψηφία και τη σημερινή αντιπολίτευση, αλλά και στη Μόσχα απευθύνεται αυτό, δεν χρειάζεται να το τονίσουμε, ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ κοντά αυτές τις ε, εκλογές. Και ε, έχουμε Ευρωπαίους και όχι μόνο παρατηρητές, τους οποίους εμπιστευόμαστε στην κρίση τους. Τώρα προσπαθεί κάποιος να θολώσει τα νερά. <laughs> Γιατί ξαφνικά έρχονται ε, από κάποια τελείως άγνωστη πηγή μια χρηματοδότηση. Ε, ε, ΜΚΟ της Φλόριδα νομίζω, της αντιπολίτευσης, που ποτέ δεν έχουν κάνει παρακολούθηση εκλογών και ξαφνικά εμφανίζονται στο προσκήνιο. μηχανίστε ή και λένε τι θα σας πούμε εμείς τώρα, τι έγινε. Και εκεί χρειάζεται προσοχή. Έχουμε την ΟΝΤΙΡ του ΟΑΣΕ, ε, θα έχουμε και παρατηρητές υποθέτω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτούς να ακούσουμε ως παρατηρητές εκλογών. Και την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, ναι, αλλά αυτοί ασχολούνται με αμυντικά ζητήματα. Και NDI και από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτοί είναι οι αξιόπιστοι που γνωρίζουν από παρακολούθηση εκλογών. Αυτούς θα πρέπει να ακούσουμε και να αγνοήσουμε κάποιους που προσπαθούν να θολώσουν τα νερά, γιατί ε, μάλλον ε, μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για τον Αγκόρνο Καραμπάχ μακάρι να είχα απάντηση. Έγινε μια συνεδρία στο Καζάν και υπήρξε αμυδρά μια ελπίδα έκφαση. Τότε ο πρόεδρος Μετβιέντεφ προσπαθούσε ενδεχομένω κάτι να κάνει καλό, αλλά απέτυχε στην τελευταία λεξούλα με την τελευταία μικροαλλαγή. Από το Καζάν και μετά δεν μεσολάβησαν πολλά και εντείνεται η πίεση και ε, ε, μετά και της Ουγγρο-Αζερικής κατάστασης που είναι πολύ μυστήρια από πολλούς ε, τρόπους, με πολλούς τρόπους. Προσπαθείτε τώρα με διπλωματικό τρόπο να κατευναστούν τα πνεύματα γιατί όταν κλιμακώνεται η κατάσταση ε, ξεφεύγει από κάθε έλεγχο με απρόβλεπτες συνέπειες. Με ηρεμία να γίνουν τα πράγματα και αυτό το λέμε και στους Αμερικανούς και στους Ρώσους που θα πρέπει να βοηθήσουν και νομίζω ότι βοηθούν και οι δύο. Και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα επανεκκίνησης της διαδικασίας που απέτυχε στο Καζάν και αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι. Δεν νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να εμπλακούμε με τέτοιο τρόπο ε, ώστε να ε, προωθούμε κάποιες πρωτοβουλίες. Όχι, να υποστηρίζουμε ε, και να διευκολύνουμε, αν θέλετε, την πολιτική διαδικασία. Γιατί όσο διανύζεται η κατάσταση, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται και εκρηκτική. Για την υπερνηστερία, θα το πω στους, αν τα λέω στους Ρώσους, ναι, με σαφήνεια, με επιμονή. Ε, σε τελική ανάλυση μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς για την Τουρκία. Και βέβαια είναι ε, εξέχον εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία. Καμιά φορά συνηθίζω να λέω ότι έχουμε δέκα στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, έτσι επίσημα. Την Κίνα, σήμερα διεξάγεται και η Σύνοδος Κορυφής αλλά κατά την άποψή μου και από την πρακτική μου εμπειρία, γιατί έχω εργαστεί στην ευρωπαϊκή εξωτερική ε, πολιτική, οι δύο χώρες με τις οποίες πραγματικά συνεργαζόμαστε ως εταίρια ε, ε, δεν χρειάζεται να το τονίσουμε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το δύο είναι η Τουρκία. Αυτό έχει να κάνει και με τη γεωγραφική του θέση. Είναι ε, τέρος κλειδί. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία και πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε καν δεν συμφωνεί η Τουρκία και συμμετέχει. Ε, ε, η διαίρεση της Κύπρου είναι δεδομένη. είχα πάει πρόσφατα και επισκέφτηκα και τις δυνάμεις των ΗΠΑ και πήγα και στην πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Βεβαίως έχουμε μια πρωτεύουσα κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαιρείται ε, όχι ε, ε, όπως είδα στο Βερολίνο από μια γραμμή και ένα τείχος, αλλά εδώ έχουμε πράσινη ζώνη, ουδέτερη ζώνη αρκετά ε, ευρεία. Ε, και αυτό θεωρείται και πολιτική και διπλωματική αποτυχία όλων των ενεχομένων. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πάρα πολύ λίγα για να μην πω τίποτα και αυτό πραγματικά μας απογοητεύει. Κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν και πρέπει να είναι πιο ενεργοί για να ξεπεραστεί ε, η διαίρεση ε, του νησιού. Αυτό είναι προς όφελος όλων και της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χώρας που ενέχεται. Καμιά φορά τίνουμε να το λησμονούμε, αλλά θα πρέπει να το τονίζουμε. Ο κύριος Πέτερ λέει είπε διάφορα πράγματα. Μερικοί από εμά ίσως να έχουμε ασχοληθεί υπερβολικά με τη Βαλκανική Χερσόνησο τα τελευταία χρόνια. Καμιά φορά έχει κάνει την αίσθηση και ότι ορισμένες χώρες έχουν κουραστεί. Υπάρχει μια κόπωση βαλκανική που έχει επέλθει. Αλλά είναι θέμα της ε, ατζέντα μας για την ασφάλεια και την ειρήνη. Δεν πρέπει να είμαστε κινδυνολόγοι και να λέμε θα ξεσπάσει πάλι πόλεμος. Δεν ξέρω, η ιστορία χρειάζεται πολύ χρόνο ε, για να ξεπεραστούν οι εντάσεις και το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να το λύσουμε είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Βοσνία μπορεί να είναι ένας τόπος που γυρνά μεγάλες απογοητεύσεις. Ε, τώρα δεν κατάφεραν να βρουν λεφτά για το Εθνικό Μουσείο του Σαράγεβο. Αυτή είναι, να ε, δείτε, δηλαδή, απογοήτευση. Ε, δώσαμε πολλά χρήματα και Σουηδών φορολογουμένων για να το ανακαινήσουμε το κτίριο. Και εγώ ήμουνα στις πρώτες ε, συνεδριάσεις ε, και καταφέραμε για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο να φέρουμε κοντά τους ηγέτες των τριών πλευρών και μπορέσαμε να το κάνουμε στο Εθνικό Μουσείο γιατί θεωρήθηκε ουδέτερη ζώνη πάνω κάτω. Αλλά τώρα δεν έχουν κονδύλια και θα κλείσει λέει το Εθνικό Μουσείο της Βοσνίας. Αυτό δεν είναι πολύ καλό ιονός για το βοσνιακό πολιτικό σύστημα. Τούτο λεχθέντο πιστεύω ότι κάνει πρόοδο η χώρα σε ανθρώπινο επίπεδο, διαπροσωπικό. Μιλήσαμε για τη διαίρεση της Κύπρου. Εκεί ε, να, δείτε διαίρεση. Στην Κύπρο βέβαια φαίνεται η πράσινη γραμμή και είναι ορατή, αλλά στη Βοσνία... Ε, κυκλοφορεί ο κόσμος, ε, δεν βλέπει τη διαίρεση. Ε, εγώ το βλέπω και η Άννα η Μπρισάντης το βλέπει γιατί είμαστε ειδικοί και έχουμε ζήσει. Αλλά πρέπει να έχει ζήσει πάρα πολύ αυτόν τον κόσμο για να βλέπει που είναι οι διαχωριστικές γραμμές. Ο κόσμο κυκλοφορεί ελεύθερα και υπάρχει διάδραση, υπάρχουν και θετικά και θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε. Μακεδονία Φιρόμ, ναι, βεβαίω χρειάζεται πρόοδο και σε αυτό. Γνωρίζω ότι ο Επίτροπος Φίλε είναι αφοσιωμένος στο να προωθήσει αυτό το θέμα και από πλευρά Συμβουλίου εμείς είμαστε διατεθειμένοι να του δώσουμε ό,τι βοήθεια χρειάζεται και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά μπορεί να μην απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις, τουλάχιστον σε μερικές και λίγα σχόλια. Είναι τεράστιο το θέμα και ε, αυτά που αποσχολούν τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τούτη τη συζήτηση στις 2.30 στην αίθουσα 5G2 με τον κάρβελτ και θα συζητήσουμε ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ειρηνή. Είστε όλοι προσκεκλημένοι για τη συζήτηση αυτή στις 2.30. Συνέφησα 5G2. Καλή σας όρεξη.